καταπολεμήσουμε την ασθένεια αυτή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα, σε ευχαριστώ, Επίτροπε κυρία Τελή. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση του θέματο. Το επόμενο σήμερα τη ημερησία είναι η παρουσία τη ακολούθηση του κυρίου Ένρικο Γερέδο Σαλόμ για τι επιπτώσει παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σε αναπτυσσόμενε χώρε και την αναπτυξιακή συνεργασία. Συνάδελφε Σαλόμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η χρηματοπιστωτική κρίση, η οικονομική κρίση ε, δημιουργεί πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις αναδυόμενες χώρες, κυρίως για τις χώρες εκείνες που έχουν χαμηλό εισόδημα. Αυτή η κρίση ε, μείωσε την ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταμάτησε σε πολλές από αυτές τις χώρες, τη μικρή ανάπτυξη που είχαν αυτές οι χώρες την τελευταία δεκαετία. Με μια μικρή ανάπτυξη μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε εξυγένση των λογαριασμών, μειώνοντας το εξωτερικό χρέος, επεκτείνοντας τις εμπορικές δραστηριότητες και με τον τρόπο αυτό είχαν περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια οι αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως, πριν από την κρίση, οι χώρες αυτές υπέφεραν πρώτα απ' όλα από την επισητιστική κρίση που έθεσε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη πάρα πολλών ανθρώπων. Έπειτα είχαμε την ενεργειακή κρίση που επίσης τους έκανε να χάσουν πολλά χρήματα γιατί τα στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, χώρες που δεν είχαν έπειτα. Κλιματική κρίση που είχε σαν αποτέλεσμα κακές οδιές κάτι το οποίο ζημίωσε ακόμα περισσότερο τις πιο φτωχές χώρες. Και επιτύχαμε και την οικονομική κρίση, η οποία προσθέθηκε στην δύσκολη κατάσταση που ήδη βρισκόντουσαν. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε, δίνοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες, ε, είπε μάλλον ότι βρίσκονταν στο τρίτο κύμα της κρίσης και είπε ότι αυτές οι πιο φτωχές χώρες υποφέρουν ακόμα περισσότερο από την οικονομική κρίση γιατί έχουν συγχρόνως και αναπτυξιακή κρίση και ανθρωπιστική κρίση και αναπτυξιακή. Όλοι οι τομείς ανάπτυξης των χωρών αυτών επλήγησαν. Η οικονομική τους ανάπτυξη που θα είναι μικρότερη το 2009 από τις προηγούμενες χρονιές περιορίστηκε το εμπόριό τους. Κάτι το οποίο πλήττει και το ισοζύγιο τρέχον λογαριασμό των χωρών αυτών. Με λιγότερες επενδύσεις από το εξωτερικό και με λιγότερη πρόσβαση στα... σε οικονομικούς πόρους. Από την άλλη μεριά, μειώθηκαν και τα εμβάσματα των μεταναστών και η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι προστέθηκαν στον κατάλογο των πιο φτωχών και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα πεθάνουν νωρίτερα σε μέρη όπως είναι η Αφρική. Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα πρέπει να ακουστεί η ευρωπαϊκή φωνή και πρέπει να ζητήσει να τηρήσουμε τις υποχρώσεις που έχουμε αναλάβει για την αναπτυξιακή μας βοήθεια προς τις χώρες αυτές και να βρούμε και νέες πηγές πόρων, επιπλέον πόρους δηλαδή, για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Πρέπει να ζητήσουμε ανακούφιση των ε, χρημάτων που πληρώνουν οι μετανάστες για τα εμβάσματα. Να μην υπάρχουν επίσης προστατευτικές ε, πρακτικές από την πλευρά μας. Και αυτό να το φροντίσουμε στον κύριο της Δόχα. Επίσης να συνεχίσουμε να καταπολεμάμε τους φορολογικούς παραδείσους και να δουλέψουμε προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία για το χρέος των πιο φτωχών χωρών. Ως εισηγητής της έκθεσης αυτής θέλησα να πετύχω ευρεία συνένεση και δέχτηκα τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αύριο όμως είμαι διατεθειμένος να υποβάλω και μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 34 της έκθεσης αυτής με στόχο να πετύχω ακόμα περισσότερες ψήφους και περισσότερη βούληση για κάτι που θεωρώ αναγκαίο, που είναι να ακουστεί δυνατά και ενωμένα η φωνή της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Ντάλι έχει το λόγο για να παρουσιάσει την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την τόσο πλήρη έκθεσή του. Όπω δικαίω τονίζεται στην έκθεση αυτή, οι αναπτυσσόμενε χώρε επλήγησαν από την κρίση πολύ σκληρότερα από ό,τι περιμέναμε φυσικά. Συγκεκριμένα, ε, πλήγησαν σε πολλές φορές μείωση των εξαγωγικών ε, εισόδων, μείωση των ροών ε, κεφαλαίου, μείωση των τιμών πρώτων υλών και αυτό είχε βέβαια σημαντικές επιπτώσεις στην αναψυχιακή ενίσχυση. Πολλές αναψυχόμενες χώρες μείωσαν τις κοινωνικές δαπάνες στον ε, τομέα της διατροφής, ε, της δημόσιας υγείας και της παιδείας. Αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία και το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο απειλείται το αποτέλεσμα μέχρι το 2015, αλλά υπάρχει μια υπαναχώρηση σχετικά με την κατάσταση των τελευταίων ετών. Παρόλα τα πρώτα δείγματα μιας ε, διεθνούς ε, ανάκαμψη, οι αναπτυσσόμενε χώρε, οπωσδήποτε θα υστερήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ε, ένα ηγετικό ρόλο για να αντιμετωπίσει την κρίση στις χώρες αυτές μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, της G20 και δράσαμε γλίγορα ώστε να αναλάβουμε συγκεκριμένε ε, δεσμεύσεις για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την Κρήτη. Πέρσι την Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα μέτρα με χρονοδιάγραμμα για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η, αντίδραση, η αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά όχι μόνο την αντίδραση της Ένωσης αλλά και των κρατών μελών που συμβάλλουν στους πόρους των διεθνών χρηματοδοτικών ε, οργάνων όπως έχουν εκληθεί να το κάνουν από την ομάδα των 20, το G20. Όπως τονίζεται στην έκθεση, η Κομισιόν έχει καθορίσει και εφαρμόσει αυτή τη στιγμή πολύ συγκεκριμένο και βραχυπρόθεσμο μηχανισμό ad hoc ευελιξία για τις πιο ευάλωτες χώρες για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να διατηρήσουν τις δαπάνες κατά προτεραιότητα στον κοινωνικό τομέα. Επίσης ε, δίνονται καινούργιοι πόροι βάσει της ε, μεσοπρόθεσμης ε, έκθεσης και υποστηρίζονται μέσα στα πλαίσια συνήθων μέσων ευελιξίας, front-loading κλπ. Η επίσημη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπαιξε και θα παίζει συνεχώς ένα σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν την κρίση. Η Κομισιόν υποστηρίζει γι' αυτό την ε, υποστήριξή σας και καλεί τα κράτη-μέλη να παραμείνουν δεσμευμένοι ούτως ώστε μέχρι το 2015 να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί. Και άλλοι δωρητές ε, θα πρέπει να καθορίσουν αυτούς τους υψηλούς ε, στόχους της αναπτυσσόμενης χώρας. Τους καλούμε όλους να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα της κρίσης των κεφαλαίων. Η Κομισιόν προσεχώς θα δημοσιεύσει μια δέσμη μέτρων ανάπτυξης για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, μια δέσμη που θα συμπεριλαμβάνει πλήρη προσέγγιση και χρηματοδότηση για επιταχυμένη πρόοδο για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης θα προβλέπεται σημαντική ενίσχυση συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνει προσκολλημένη στη δεσμεύση της η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξακολουθεί να παίζει ηγετικό ρόλο στον τομέα. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Περνάμε αμέσως στη διαδικασία Κατσουδιάη. Η συνάδελφος Βασέσκου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η οικονομική και δημοσιονομική κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ την Μολδαβία, που είναι αναδιόμενη χώρα. Η οικονομία της χώρας αυτής έχει μειωθεί 9% πέρυσι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 6% έχει ανέβει ανεργία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν επενδύσεις στη χώρα αυτή. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει ζητήσει από εννέα συμβούλους που τους έχει προσλάβει για ένα χρόνο να βοηθήσουν ε, τα αρμόδια υπουργεία. Οι Ρουμάνοι και οι Μολδαβοί μιλάμε την ίδια γλώσσα, οπότε οι Μολδαβοί μπορούν να έχουν βοήθεια από εμάς σε όλους τους τομείς. Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε ε, με τα εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες Μολδαβοί στην Μολδαβία και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη χώρα. Χαίρομαι λοιπόν που η Μολδαβία είχε 2,6 ενίσχυση για την περίοδο 2011 με 2013. Ο Πρωθυπουργό της Μολδαβίας κατάφερε να πετύχει αυτό το ποσό σήμερα στη διάσκεψη των δωρητών. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την κρίση, αυτοί που επλήγησαν περισσότερο είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Με τις αβεβαιότητες, με το διεθνές εμπόριο που έχει μειωθεί, με τους μετανάστες που έχουν αυξηθεί, όλα αυτά αποτελούν συμπτώματα μιας κρίσης που έχει προκληθεί και έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Εμείς ζητήσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υπολογίσει τη ζημιά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό θα γίνει εν ώψη της διάσκεψης των 20. Γι' αυτό και προτείναμε να υπάρξει ένας φόρος για τις τραπεζικές συναλλαγές, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες αυτές. Χαίρομαι που ο κύριος Γερέρο έχει δεχτεί τις προτάσεις αυτές και τον συγχαίρω για την εξαίρετη εργασία του. Σας ευχαριστώ, συνάδελφο. Σμίτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αργά είναι, τέτοια ώρα. Θα σα απευθύνω χαιρετισμού και σε εσά και συγχαρητήρια στον εισηγητή. πιστεύω ότι αυτή η κρίση θα ξεπεραστεί με περισσότερο ελεύθερο εμπόριο και παγκοσμιοποίηση, όχι προστατευτισμό. Θα πρέπει η Ευρώπη να κρατήσει τι αγορές αγορέ ανοιχτέ για να περάσει αυτή την ύφεση και να προσπαθήσει να καταπολεμήσει και τη φτώχεια μέσω ανοιχτή προσέγγιση. Σε λίγε μέρε η Ισομερή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ευρωπαϊκή Ενώση συναντηθεί στην Τενερίφη και οι συνάδελφοι των χωρών και πάντα αναφερόνται τα προβλήματα που δημιουργούνται από επιδοτούμενα αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκή Ενώση που καταφθάνουν σε αγορέ του. Η πολιτική, η πολιτική μας αφορά τη δημιουργία υγιών αγορών για γεωργικά προϊόντα στις χώρες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγηθεί λέει η Επίτροπος. Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Χρειάζεται δίκαιο εμπόριο, fair trade κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι κρίσεις που αναφέρονται στην έκθεση, η επισητιστική, η ενεργειακή, η κλιματική, η οικονομική και η κοινωνική, αποτελούν συμπτώματα της διαρθρωτικής κρίσης η οποία μας πλήττει εδώ και δεκαετίες κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική αλλά και άλλες περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών αυτών, αλλά υπάρχει κάτι κοινό, ότι μειώνονται οι εξαγωγές τους, ε, πέφτουν οι τιμές των πρώτων υλών τους, Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση της γεωργίας και η επιρροή των ξένων χωρών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι χώρες αυτές λοιπόν είναι θύματα εκβιασμού, κυρίως όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές τους. Και έτσι οι χώρες αυτές είναι εξαρτώμενες και έχουν όλο και λιγότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που χάνουν πόρους. Το χρέος τους έχει φτάσει σε τεράστια επίπεδα και η εκμετάλλευση των χωρών αυτών συνεχίζεται με όλο και υψηλότερα επίπεδα. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφα. Είναι θέμα δικαιοσύνης επίσης να τηρείτε το χρόνο γόρευσης. Τελευταίος ομιλητής για το ΚΑΤΣΔΙΑΗ. Συνάδελφος μιλούσαν ένα λεπτό το πολύ. Η μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση από τη δεκαετία του 30 της περισμένης δεκαετίας δεν έπληξε μόνο την Ευρώπη. Οι αναψώμες χώρες υποφέρουν ιδιαίτερα. Και είναι η κρίση που φταίνε το λιγότερο. Κερδοσκοπία που θέλει ψηλά κέρδα, ιδίω στον σαξονικό κόσμο, οδήγησαν τον κόσμο στα πρόθυρα της ε, οικονομικής καταστροφής. Ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν τεράστια χρέη στα κράτη για να μπορέσει να υπάρχει μια ανάκαψη της οικονομίας, αυτό η άγουσα δεν είναι δυνατή σε αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν μπορούν να ενδυναμώσουν μόνες τους τις ε, οικονομίες τους. Ε, πρέπει να αμυνθούν κατά των εισαγωγμένων προϊόντων που ρίχνονται στην αγορά και που υποσκάπτουν την εσωτερική τους οικονομία. Η κλασική αναπτυστική βοήθεια μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποτύχει. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί το πρόβλημα στην ρίζα του, να παγωρευτούν οι κερδοσκοπείς και να εισαχθεί ο φόρος για τις κεφαλικές συναλλαγές. Πρώτος ευχαριστώ στον Μόλτσερ. Θέλει η το λόγο. Φαίνεται ότι όχι. Οπότε ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματο. Η ψηφοφορία γίνεται αύριο. Η επόμενη συνεδρίαση είναι αύριο, 5η 25 Μαρτίου 2010, 9 με 1 το πρωί. Έχει δημοσιευτεί η ημερησία διάταξη. Μπορείτε να τη διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, να του ευχαριστήσω που ήταν εδώ και επίση του συνοδεύουν.